So, dear colleagues, good morning. Um, Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Ακόμα και αν είναι πολύ λίγα τα μέλη ε, παρόντα στην αίθουσα, να αρχίσουμε παρακαλώ. Θα συνεχίσω γερμανικά. Um, unser Punkt jetzt, Nummer 10 ε, Σημείο 10 11 δηλαδή, Γενικό Προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το Οικονομικό Έτο 2018. Ο Μόρτεν Λόκεγκαρτ είναι ο εισηγητή μα. Στι 30 Μαου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε και δημοσίευσε το σχέδιο προϋπολογισμού ε, και σας έχουν ε, σταλεί ε, όλα τα έγγραφα. Υπάρχει ένα σημείωμα της γραμματείας για την Επιτροπή μας σε ό,τι αφορά τις δικές μας γραμμές και θέσεις του προπολογισμού δύο βασικά τμήματα της διαδικασίας του προπολογισμού υπάρχουν. Από τη μια γνωμοδότηση ε, για το σχέδιο προπολογισμού που πρέπει να κατατεθεί στις 29 έκτου και ε, η αλλαγή του σχεδίου τροποποίηση ίδια. Σήμερα θα κάνει τις προτάσεις ο κύριος Λόκεγκαρτ και πριν του δώσω το λόγο θέλω να σας θυμίσω ότι Πρώτον, προθεσμία για την ε, κατάθεση των τροπολογιών στον προπολογισμό στην Επιτροπή μας λήγει στις 26 Ιουνίου στις 6 ώρα το απόγευμα. Τη Δευτέρα είναι. Και οι συντονιστές στις 22 Μαρτίου αποφάσισαν οι τροπολογίες να ε, υποβάλλονται στα αγγλικά παρακαλώ. Και τρίτον, πρόταση για πιλωτικά προγράμματα ή προπαρασκευαστικές δράσεις ε, οφείλουν να υποβάλλονται ως τροποποιήσεις του προϋπολογισμού. Αυτά εισαγωγικά θα δώσω μέσα στο λόγο στον Μόρτεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Δύο λόγια μόνο για τη θέση Επιτροπής Προϋπολογισμού, για το σχέδιο Γενικού Προϋπολογισμού του 2018. Θα γνωρίζετε οι περισσότεροι τη γενική μου θέση. Έχω καταθέσει πριν από λίγες εβδομάδε τη γνώμη μου για το τριμερή διάλογο. Έκτοτε είχα την ευκαιρία να συζητήσουμε περισσότερους και τους δικούς μας εμπειρογνώμονε για τον προπολογισμό της Επιτροπής Πολιτισμού για τα βασικά διαδικαστικά θέματα. Σε αντίθεση με τον περασμένο γύρο συζητήσεων που δεν ξέραμε τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακόμα, σήμερα τη γνωρίζουμε. Όπω είπε και η κυρία Τρίπελ, Έχουμε τα στοιχεία, τα αριθμητικά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να τονίσω τα σημαντικότερα θέματα. Πρώτον, λυπούμαστε βαθιά ακόμα που δεν έχουν προσθέσει τα 50 εκατομμύρια που είχαν προσημειωθεί για το Erasmus Plus στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο μέχρι το 2020. Εάν δεν μπορούμε να βρούμε τα 50 εκατομμύρια σε μία δόση, τουλάχιστον σε τρεις δόσεις, το 18 α πούμε, την πρώτη δόση 18, για να μπορεί το πρόγραμμα Εράσμου να λειτουργεί πλήρως. Δεύτερον, ανησυχούμε για τον προπολογισμό σε ό,τι αφορά το σώμα αλληλεγγύης ε, το οποίο επιβαρύνει το Erasmus Plus και θέλουμε να μας τα διευκρινίσει αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδιαίτερα πώς θα συνδεθεί αυτό το νέο σώμα με ε, την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία. 18 εκατομμύρια ευρώ νέο χρήμα έχουν ε, μπει στην άκρη για το θελοντικό σώμα, αλλά παρακαλώ αυτά να μην τα πάρουν από το Erasmus Plus. Και είμαι πολύ περίεργος να ακούσω τι θα πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τρίτον, υπάρχει μια χρόνια υποχρηματοδότηση των προγραμμάτων μας, του Creative Europe και άλλων πολιτιστικών προγραμμάτων. Εμείς ζητούμε αύξηση φυσικά των κονδυλίων και λυπούμεθα για το γεγονό ότι υπάρχει περικοπή 740.000 ε, ευρώ. Βέβαια δεν είναι πάντα ε, μεγάλη απορρόφηση τα θετικά. Ε, έχουμε το Creative Europe για να χρηματοδοτήσουμε το 2018 που είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Θέλουμε όμως ξεχωριστή γραμμή και θέση στον προπολογισμό για τα 7 εκατομμύρια ε, που έχει δεσμευτεί το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πάντα για αυτή τη χρονιά. Αυτό το τέταρτο, πέμπτο. Υπάρχουν ε, δράσεις για τα multimedia και εδώ είναι υποχρηματοδοτούμενο το μέτρο. Θα πρέπει να βρεθεί μια μακροπρόθεσμη ε, λύση για το Euronet Plus, να συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα συνεργασίας των ραδιοφώνων με σωστό χρηματοδοτικό πλαίσιο ε, και αυτό να φαίνεται στον προϋπολογισμό. Ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για να υπάρξει βιωσιμότητα του Euronet και μετά το 2018. Είναι πολύ καλοδοκιμασμένο πανευρωπαϊκό ραδιοφωνικό δίκτυο το Euronet. Θα πρέπει να τονίσουμε την αξία αυτών των προγραμμάτων ε, Το New Narrative for Europe, ένα νέο φύγημα για την Ευρώπη, είναι κάτι το οποίο προσελκύει νέους και ζητούμε να συνεχιστεί αυτή η πρωτοβουλία μέσω του Erasmus+. Έβδομα, ο αθλητισμός επίσης είναι πολύ προσφυλές θέμα για μας και μάλιστα ο, όχι ο πρωταθλητισμός, ο καθημερινός αθλητισμός των πολιτών και προάγει τις ευρωπαϊκές αξίες. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχουν δράσεις εκεί, γι' αυτό καλωσορίζουμε την απόφαση να συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 2017 ένα κονδύλι για ειδικά ε, αθλητικά γεγονότα και διοργανώσεις ετήσια και ζητήσαμε ένα εκατομμύριο. Τώρα για το 2018 θα πρέπει να προ Άγουμε και να τονίσουμε τη σημασία του αθλητισμού και της άσκησης ε, των πολιτών. 3.000 είναι εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί στα διάφορα κράτη-μέλη με πάνω από 1,5 εκατομμύριο συμμετέχοντες. Ε, όλα αυτά συνάδουν με την τελευταία μας γνωμοδότηση που υποστηρίξατε πολλοί από εσά σε μεγάλο βαθμό και ελπίζω γρήγορα να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Προσβλέπω στη συνεργασία, στη συζήτηση και στη συμμετοχή σας. Η ταχύα αντίδραση είναι βεβαίω απαραίτητη. Ε, θέλω να σας θυμίσω, όπως είπε και η Πρόεδρος, ότι έχουμε προθεσμία για τις ε, τροπολογίες κοντινή σε λίγες μέρες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Okay, thank you, Morgan, And now I would uh, like... Ευχαριστώ, Μόργαν. Σκιώδε τώρα να πάρουν το λόγο. Ο κύριο Τσαβίσκη, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν πρόκειται να επαναλάβω τη συζήτηση που έχουμε ήδη κάνει επανειλημμένα. Απλώς ε, θα χάναμε χρόνο εάν το έκανα. Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε σύντομοι. Πρέπει οπωσδήποτε να θυμίσουμε ότι αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι το Erasmus Plus ε, και ε, πιστεύουμε ότι είναι περιορισμένη η χρηματοδότηση σε σχέση με τα 50 εκατομμύρια που θα πάνε στο σώμα αλληλεγγύης. Το Erasmus Plus ε, είναι, μάλλον από το Erasmus Plus ωφελείται το σύνολο των νέων, ενώ το σώμα αλληλεγγύης είναι κάτι πολύ πιο ειδικό ε, και ε, αφορά ένα πολύ συγκεκριμένο αριθμό ε, ατόμων και δραστηριοτήτων. Αυτό που είναι λοιπόν σημαντικό τώρα και θα είναι πιο σημαντικό και σε λίγους μήνες είναι το Erasmus Plus. Επίσης ε, πιστεύω ότι έχουμε επιφυλάξεις στην Επιτροπή μας γιατί ε, τελικά τα ποσά επί των θεμάτων που είχαμε εμεί θέσει ως προτεραιότητες είναι πάρα πολύ ε, περιορισμένα και επίσης υπάρχει και περισσότερος αριθμός νέων ε, προτεραιοτήτων και πρωτοβουλειών. Ε, ο συνέργος αναφέρθηκε σε κάποια σημεία σημαντικά. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπεραμεινθούμε στεναρά των θέσεών μας. Έρασμους ε, Πλάς, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ραδιοφώνων, αυτά είναι πολύ σημαντικά για μας. Επίσης ε, το εμπόριο έργων τέχνης, ε, γνώση ε, ε, περί, την, τον πολιτισμό. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να επιτύχουμε αυτά τα επιπλέον 4 εκατομμύρια και για την πολιτιστική κληρονομιά. Εν πάση περιπτώσει, τα ποσά είναι πολύ μικρά ούτως ή άλλως και και νομίζω ότι και για το Creative Europe ε, ε, θα τα χρειαζόμαστε έτσι κι αλλιώς τα επόμενα χρόνια ε, και μέχρι το 2019 μας είχαν υποσχεθεί ότι θα δοθούν τα 4 εκατομμύρια στην Creative Europe και αν δεν δοθούν θα πρέπει να βρεθούν άλλες πηγές χρηματοδότησης και οπωσδήποτε θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι οποιαδήποτε επιπλέον κονδύλια ε, θα αφορούν την Creative Europe και θα χρηματοδοτήσουν την ε, Creative ε, Europe. Νομίζω ότι θα πρέπει να αγωνιστούμε έτσι ώστε οι θέσεις μας να περάσουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μοργάνο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για την ε, γνωμοδότηση που έκανε και για ορισμένα σημεία τα οποία ανέφερε, γιατί θεωρώ ότι αποτελούν συγκεκριμένο σημείο αναφοράς ε, για να αντιμετωπιστούν ε, θέματα προϋπολογισμού που όμως είναι πολύ σημαντικά για τον πολιτισμό, τον αθλησμό και για τους νέους. Είναι γεγονός ότι τα ποσά είναι σχετικώς χαμηλά. Αλλά αυτό είναι άμεση άμεση επίπτωση ε, το, της υποχρηματοδότησης ε, της ε, Δημιουργικής Ευρώπης και της Ευρώπης για τους πολίτες. Εγώ εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ένας τρόπος για να λυθεί το πρόβλημα αυτό είναι να δοθούν ήδη οι πόροι στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. κοιτάξτε, όσον αφορά ε, ε, το, την χρηματοδότηση, προσέξτε μόνο τη χρηματοδότηση, όχι την ουσία ε, του Σώματος Αλληλεγγύης. Έχουμε πρόβλημα με, αυτήν, με αυτή τη χρηματοδότηση. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια, μια χρηματοδότηση τέτοια που να επιτρέπει μεγαλύτερες επενδύσεις. Και άλλωστε, όπως είπε και ο εισηγητής, προβληματίζομαι γιατί Αυτά τα 50 εκατομμύρια, ε, τα πρόσθετα που είχαν υποσχεθεί ε, οι θύνοντες ε, για τον έρασμο πλάσα, δεν τα βλέπουμε. Αντιθέτως, χρηματοδοτούνται ε, τα σώματα αλληλεγγύης τα οποία είναι ε, συνδεδεμένα με τον Erasmus Plus. Εν πάση περιπτώσει επαναλαμβάνω ότι αυτά τα 50 επιπλέον εκατομμύρια που περιμέναμε δεν τα βλέπουμε. Επίσης στο σχέδιο προϋπολογισμού βλέπουμε ότι από το Erasmus Plus λείπουν ακριβώς αυτά τα 50 εκατομμύρια. Και Βεβαίως ε, οι, νέοι και οι νέοι του Erasmus Plus είναι αυτοί που υποφέρουν περισσότερο. Παραδόξως, εάν θυμηθούμε Πόσες φορές και σε διάφορα φόρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει αναφέρει ότι ε, θέλει να επενδύσει στους νέους, πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, δοθούν τα χρήματα τα οποία είχαν προβλεφθεί στον προγραμματισμό. Και λέω ότι παρότι είναι μικρός ο χρόνος υποβολής τροπολογιών, θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε απολύτως νομίζω στην Επιτροπή μας ότι θα πρέπει να υποβληθούν αυτές ε, οι τροπολογίες ε, οι οποίες θα αναφέρονται στον προϋπολογισμό ε, και που από κοινού κατά κάποιο τρόπο θα αναφέρονται στην ανάγκη να βρεθούν αυτά τα χρήματα τα υπεσχημένα. Και βεβαίως να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για την εργασία του. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μοργάνο. Θα μιλήσω εγώ ως σκιώδης των Πρασίνων για τον προπολογισμό. Αυτό που θέλω να τονίσω, να υπογραμμίσω και αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έχουμε αυτή την κατάσταση της υποχρηματοδότησης των προγραμμάτων μας, της Δημιουργικής Ευρώπης, της Ευρώπης για τους πολίτες και του Εράσμους βέβαια. Ακόμη και αν υπήρξε μια μικρή αύξηση, ξέρετε ότι δεν είναι επαρκή και θα μπορούσαν να είχαν γίνει πολύ περισσότερα πράγματα και αυτό θα ήταν πολιτικά σωστό και καλό να ε, συμπεριλαμβάνονται περισσότερο οι νέοι. Οπότε πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα δοθούν αυτά τα 50 εκατομμύρια που μα έχουν υποσχεθεί και νομίζω ότι αυτή θα είναι η κοινή μα θέση ω Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδεία. Τώρα, να μιλήσω για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη. Όπω γνωρίζετε, στην αρχή είχα πολλέ επιφυλάξει ω προ τη χρηματοδότηση αυτού του σώματο και είχα πει ότι δεν πρέπει να πάρθουν χρήματα από το Erasmus Plus. Τώρα η Κομισιόν μα εξήγησε ότι παίρνει ε, χρήματα από το Erasmus που πάει στο σώμα ε, εθελοντισμού και ενσωματώνουν ε, το σώμα αυτό και τον προπολογισμό του σε αυτό το νέο σώμα αλληλεγγύης. Αν τα πράγματα είναι έτσι, θα μπορούσα να πω εντάξει. Ε, μπορούμε ε, να μεταφέρουμε ε, χρήματα από το σώμα αλληλεγγύης και από εκεί και πέρα αξιοποιούν 86 εκατομμύρια νέα χρήματα, φρέσκα χρήματα. Φυσικά Καλά κάνουν και τα κάνουν αυτά, αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι χρειάζεται νέα πρόσθετα χρήματα και κονδύλια. Και γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει να καλέσουμε και την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να, διατεθούν χρήματα από τα μη διατηρημένα κονδύλια. Νομίζω ότι το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε είναι ότι είναι σωστό να, ε, να χρησιμοποιηθούν μεν τα χρήματα του σώματος εθελοντισμού για το σώμα αλληλεγγύης, αλλά δεν θα πρέπει να παρθούν καθόλου άλλα χρήματα από το Erasmus ε, Plus. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε απόλυτα ποιες είναι οι δικές μας απαιτήσεις και προσδοκίες. Επίσης, συμφωνώ με αυτό που είπατε για το, για το έτος πολιτιστικής κληρονομίας, για τα πολυμέσα και τον ε, την ποιοτική δημοσιογραφία. Νομίζω ότι και σε, αυτό, σε αυτούς τους τομείς έχουμε καλά προγράμματα. Υποστηρίζω και την προσέγγιση για το Euronet Plus. Νομίζω ότι πρέπει και εκεί να αυξηθεί ο προπολογισμό, Αθλητισμός, μαζικός αθλητισμός, ενσωμάτωση ανθρώπων από ε, μειονεκτικά στρώματα του πληθυσμού, ιδίως για ε, μειονεκτούντα μάλλον ε, στρώματα του πληθυσμού, μετανάστες κτλ. Με όλα αυτά που είπατε συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι πριν ξεκινήσει η συζήτηση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει η Επιτροπή μας να έχει σαφή θέση για το τι περιμένουμε να γίνει Ιδίω για τα προγράμματα βεβαίως για τα οποία εμεί είμαστε αρμόδιοι και που είναι πολύ σημαντικά για τους πολίτες, ακριβώς γιατί βοηθούν στην, ε, στην άνοδο της αποδοχής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και σε όλα αυτά βεβαίως συμβάλλουν ο αθλητισμός, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κτλ. Αυτά ε, και ο λόγος τώρα στην Σίλβια Κώστα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τους σκιώδη για τη δουλειά τους ε, και τον εισηγητή μας. Συμφωνώ με την κυρία Τρούπελ, θα πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα ε, στο Κοινοβούλιο, πέρα από την Επιτροπή μας. Κόπτεται συνεχώς το Κοινοβούλιο για την αλληλεγγύη, για τον πολιτισμό, για τους νέους. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν μια συνέπεια. Θα πρέπει να κάνουμε πολύ σκληρή δουλειά με την Επιτροπή Προϋπολογισμών αλλά και με άλλες επιτροπές για να είναι αυτό το μήνυμα το ε, στεναρό και το ηχηρό πραγματικό. Ε, περιμένανε λέει να έχουν την ενημέρωση για το Brexit, γι' αυτό καθυστέρησαν. Ε, αυτά είναι τα επιχειρήματα και γιατί ε, δεν έχουν δοθεί τα χρήματα που έπρεπε να εγγραφούν στο κεφάλαιο Erasmus Plus. συμφωνώ επίσης με αυτά που λέτε για το σώμα αλληλεγγύης. Πρώτα πήρανε λεφτά από το Εράσμος και μετά μιλήσανε για τη νομική βάση και έχει γίνει ένα μπέρδεμα. Ε, υπάρχει σήμερα εθελοντική υπηρεσία που γίνεται εθελοντικό σώμα. Νομίζω ότι εκεί υποτιμήσαμε και υποπρικοδοτήσαμε το Creative Europe, Δημιουργική Ευρώπη. Ε, σε αυτά τα προγράμματα υπάρχουν προγράμματα που έχουν δείκτη ε, αποτελεσματικότητας ή επιτυχίας 12% μόλις. Ε, για τη δημιουργική Ευρώπη ε, θα πρέπει ε, να κάνουμε πολύ συστηματική δουλειά σε σχέση με αυτά που αποφασίστηκαν το 2015. Όλοι ξέρουμε ότι είναι προτεραιότητες αυτά τα θέματα. Το 2018 είναι έτος πολιτιστικής κληρονομιάς και το Creative ε, ε, Europe αυξάνεται λίγο. Ε, πρέπει να παρακολουθούμε όλα τα προγράμματα, όλα τα κονδύλια για να ε, μπορούμε αυτά τα πιλωτικά προγράμματα να τα εκτελούμε με σωστό τρόπο. Γιατί είναι υπέρ της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Θέλω να δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. <coughs> Euh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμα μέρη, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τη βάγια υποστήριξη στην Επιτροπή σας κάθε φορά που ερχόμαστε για τα προγράμματα και τις λύσεις. Ωστόσο θα πρέπει να ε, διευκρινίσω κάποια πράγματα ε, για τα όσα προτείνουμε στην ενδιάμεση αναθεώρηση, το περίφημο top-up για 100 εκατομμύρια για το Erasmus Το, τα 50 τα πήραμε το 2017, άρα μένουν 50 για να κατανεμηθούν στα επόμενα τρία έτη, 18, 19, 20 και είναι φυσιολογικό να εκφράζετε κάποια έκπληξη που δεν τα βλέπετε στο προπολογισμό του 2018. Γιατί όταν καταρτίστηκε το σχέδιο προπολογισμού δεν είχε ληφθεί απόφαση. Αυτή ελήφθη τη Δευτέρα ή την Τρίτη νομίζω μετά ε, τις εκλογές ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και τώρα ετοιμάζουμε μια τροποποιητική επιστολή με τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμών για να προτείνουμε τα διάφορα top-up και τις αυξήσεις όχι μόνο στο Εράσμος αλλά και σε άλλα προγράμματα που αποφασίστηκε τώρα στην αναθεώρηση. Η Γενική Διεύθυνση Παιδείας και Πολιτισμού θέλει για το 2018 να έχει διαθέσιμα τα 2018 για να το σχεδιάσουμε και για τα μελλοντικά. Γιατί ξέρετε ότι η καμπύλη αυξάνεται, έχει μια ραγδαία αύξηση στη διάρκεια του 2019 στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού προγράμματος, πρέπει να τα δούμε όλα αυτά, πλαισίου μάλλον, ε, η καλύτερη λύση δεν είναι να ε, τα μοιράσουμε στις διάφορες χρόνιες ε, αναλογικά ή αποσπασματικά. Επίσης θέλω να διευκρινίσω ότι τα 50 εκατομμύρια ζητήθηκαν και λήφθησαν για την ενίσχυση του Erasmus Plus. Δηλαδή, αν έχετε την παραμικρή αμφιβολία, είναι ακριβώς για αυτό το πρόγραμμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε να ενισχύσει τα προγράμματα που είναι επιτυχημένα, που λειτουργούν καλά και ε, που έχουν ε, χαμηλή επιτυχία. Άλλο. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατανοεί την ε, Ανησυχία σας. 197 εκατομμύρια ευρώ για τρία χρόνια βγαίνουν από το Εράσμος για να πάνε στο ΣΑΜΟ Όπως γνωρίζετε, θα έχει προπολογισμό συνολικό 341 εκατομμύρια ευρώ, αυτό προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά όπως πολύ καλά εξηγήσατε κυρία Πρόεδρε, αυτό θα πρέπει να το δούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Τι κάνουμε εμείς. Υπάρχει η εθελοντική υπηρεσία που ήταν στο Erasmus Plus. Αυτό φεύγει και μπαίνει στο εθελοντικό σώμα τώρα. Η εθελοντική θητεία βγαίνει από το Erasmus Plus και ε, υπάρχουν και νέα χρήματα και ε, συμπερίληψη άλλων κονδυλίων από άλλα προγράμματα που δεν έχουν βοηθήσει για την νεολαία. Και τελικά θα έχουμε περισσότερα χρήματα από ό,τι είχαμε στην αρχή ε, στην Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία. Δηλαδή η ιδέα είναι να προσφέρουμε 100.000 θέσεις μέχρι το 2020. Ο πρόεδρος Γιούνκερ ο ίδιος το έχει θέσει ως προτεραιότητα. Δηλαδή πολλά περισσότερα από ε, το μέσο του Erasmus Plus. Όπως γνωρίζετε το 25% είναι νέα χρήματα, άρα υπάρχει περιθώριο και ε, θα έχει και πολύ σημαντικότερο αντίκτυπο στην νεολαία. Άκουσα ανησυχίες για αυτό το θέμα της νεολαίας η οποία πλήττεται. Το αντίθετο συμβαίνει. Ενισχύσαμε τις προσπάθειες που κάνουμε για τη νεολαία. Αυτά είναι τα δύο θέματα που θα ήθελα να ε, ξεκαθαρίσω. Ευχαριστώ. Ο λόγος και πάλι στον κύριο και στη συνέχεια στον κύριο Μόργαν και μετά στον εισηγητή μας. Ευχαριστώ πολύ με ανησυχούν λίγο οι πληροφορίες που μας δόθηκαν μόλις. Να μην ξεχνούμε ότι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ε, δεν ε, ε, τελειώνει την, την, τη λειτουργία του ούτε φέτος ούτε του χρόνου. Υπάρχουν ε, χρήματα που προβλέπονται και μάλιστα σημαντικά ποσά που προβλέπονται και για το 2019 και για το 2020. Επίσης, όλα αυτά τα χρόνια θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί και η Δημιουργική Ευρώπη και όλα αυτά τα χρήματα έρχονται από, προέρχονται από τον ίδιο Κορβανά. Και φαίνεται ότι θα γίνει αυτό εις βάρος του Erasmus Plus. Τι θέλω να πω, δεν μπορούμε να, να έχουμε στο επίκεντρο τη προσοχή μα μόνο την επόμενη χρονιά, το 2018. Υπάρχει ένα πιο μακροπρόθεσμος σχεδιασμό που πρέπει να έχουμε υπόψη μα και δεν θέλουμε να δημιουργηθούν ε, ελλείψει ε, χρηματοδοτικέ όσον αφορά το Erasmus Plus. Όσον αφορά τα ε, έγγραφα που περιγράφουν τι μελλοντικέ προοπτικέ, υπάρχει το σχέδιο προπολογισμού το, ο, ο υλοποιηθής προϋπολογισμός των προηγούμενων ε, ετών και όλα αυτά μπορούν να μας οδηγήσουν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Αυτό που πρέπει σε σχέση με το Erasmus Plus πρέπει οι πληρωμές να συνεχίσουν να καταβάλλονται ομαλά, χωρίς ε, κενά ε, και χωρίς διακοπές. Ευχαριστώ κύριος Μόργαν. Κοιτάξτε, υπάρχει κάτι το οποίο δεν μπορώ να το καταλάβω σε σχέση με την θέση που εξέθεσε η Κομισιόν. Υπάρχει μία ανακοίνωση της 30 Μαΐου που λέει ότι η πρόταση προπολογισμού για το 2018 έχει γίνει ε, σαν να είχε εγκριθεί ήδη η ε, αναθεώρηση. Επομένως, από τη στιγμή που εγώ διαπιστώνω ότι στο προσχέδιο προπολογισμού λείπουν 50 εκατομμύρια του Erasmus Plus. Δεν είναι δυνατόν να, ε, να ε, προσυπογράψω, επομένως, ε, άρα τα πράγματα δεν πάνε καλά. Επομένως, πρέπει να πω ότι το πλαίσιο το οποίο αναφέρατε δεν ισχύει ανακοίνωση της 30 η Μαΐου. Λέγεται, αναφέρεται ότι ε, η πρόταση του προπολογισμού γίνεται λες και είχε εγκριθεί ε, η ε, πρόταση. Και γιατί λείπουν λοιπόν στην πρόταση προϋπολογισμού, γιατί λείπουν τα 50 εκατομμύρια. Δεν είναι λογικό. Modern, oh, sorry. It was a direct question to the Commission. Αυτή ήταν, λέει η Πρόεδρος, άμεση ερώτηση στην Κομισιόν. Μπορείτε να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι κάτι δεν έγινε καλά κατανοητό. Τη στιγμή που που προετοιμάστηκε ο προπολογισμό, τα 50 εκατομμύρια ε, είχαν μπλοκαριστεί εν αναμονή των εκλογών ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένω, είχαν μπλοκαριστεί, δεν περιλαμβάνονται τα 50 εκατομμύρια ε, ούτε για το Erasmus Plus ούτε για πουθενά αλλού. Τώρα που ξεμπλοκαρίστηκαν, α πούμε, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο θα μπουν και τα χρήματα αυτά στον προπολογισμό και θα ανάλογα με τα περιθώρια τα οποία ε, ε, υπάρχουν και ανάλογα ε, και με τα όρια των δημοσιονομικών αρχών θα, θα μπουν τα χρήματα αυτά ανά προγράμματα. Είναι το δεύτερο τμήμα λοιπόν του top το οποίο δεν έχει περιληφθεί το τμήμα 18-20, 2018 μέχρι 2020, ε, δεν είχε προϋπολογιστεί, μάλλον δεν είχε συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό. Θα ληφθεί η επίσημη απόφαση στο Συμβούλιο όσον Okay, then we will hope that... Ωραία, επομένως ε, ελπίζουμε ότι θα αντιμετωπιστεί το θέμα, ευελπιστούμε δε ότι θα αντιμετωπιστεί θετικά ε, και όταν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της αναθεώρησης ε, των MFF, τότε θα ε, λυθεί και το ζήτημα. Μόργαν, σου δίνω ξανά τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι η συζήτηση που μόλις ε, έλαβε χώρα απεικονίζει ακριβώς την κατάσταση, δηλαδή ότι κάποια ζητήματα χρήζουν περαιτέρω συζητήσεως. Και ως εισηγητής ε, το λέω αυτό, ε, ότι χρειάζομαι ε, και κάποιες άλλες απαντήσεις σε ερωτήσεις μου από πλευρά τη Κομισιόν. Ελπίζω ότι μπορούμε να κανονίσουμε έτσι μια συνάντηση έτσι ώστε να διευκρινιστούν όλα τα σημεία γιατί ακόμα υπάρχουν κάποια που χρήσουν διευκρινήσεως. Βεβαίω ευελπιστώ ότι οι τροπολογίε των συναδέλφων ε, θα αναφέρονται ακριβώ σε αυτά τα προβλήματα έτσι ώστε τουλάχιστον από τη δική μας ε, Επιτροπή να ε, είναι σαφής η θέση και νομίζω, αν ερμηνεύω σωστά τα σχόλια που άκουσα σήμερα, ε, νομίζω ότι οι τροπολογίες οι οποίες θα υποβληθούν θα είναι σε αυτή τη γραμμή, γιατί έχουμε δηλαδή κοινή κατανόηση των ε, θεμάτων και ότι είμαστε μαζί σε αυτό το ζήτημα. Θα συνεχίσω με την, ε, επί τη αυτής της κοινή κατανόησης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Περιμένω λοιπόν στις επόμενες μέρες τις τροπολογίες σας και μετά θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. And, uh, let me remind... Ευχαριστώ Μόργαν. Να σας πω για μία ακόμα φορά. Δευτέρα 26 του μηνό στις 6 το απόγευμα λίγη η προθεσμία υποβολής των τροπολογιών. Ε, επόμενο σημείο 11 της ημερησίας διατάξεως στα γερμανικά. Μιλάμε για την ε, γνωμοδότηση, για την έκθεση ε, πρωτοβουλίες της Επιτροπής ε, Απασχόλησης για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τους ανθρώπους με αναπηρίες. Συντάκτια τη γνωμοδότησης είναι η Julie Ward. Την, ε, τον Φεβρουάριο του 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ενδιάμεση έκθεσή της για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα άτομα με αναπηρίες. Αυτή η στρατηγική είναι το βασικό μέσο για την υποστήριξη της υλοποίησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στόχοι της στρατηγικής ε, χωρίζονται σε 8 τομείς, μεταξύ αυτών και ε, η εκπαίδευση και η κατάρτιση. Η χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και διαβίου μάθησης έχει ως σκοπό να βελτιώσει τις ευκαιρίες και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων με αναπηρίες. Σε αυτό, τον, ε, σε αυτό το πλαίσιο το Erasmus Plus διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο γιατί διευκολύνει την κινητικότητα για τους, τα άτομα με αναπηρίες. Η συγκίτριά μας, Julie Ward, λοιπόν, έχει ασχοληθεί εκτενώς με αυτά τα θέματα και γι' αυτό μπορεί να μας, θα μας παρουσιάσει τώρα πού μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα. Πρωτού δώσω το λόγο στην Τζούλη, να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι 29 Ιουνίου στις 2 το μεσημέρι. Επίσης να σας επισημάνω ότι η συζήτηση, η ψηφοφορία που θα γινόταν στις 28 Σεπτεμβρίου θα γίνει στις 10 Οκτωβρίου τελικά. Ευχαριστώ πολύ, ε, Τζούλη. Ευχαριστώ. Με μεγάλη χαρά ανέλαβα αυτό το θέμα γιατί ασχολούμαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια ε, με τα θέματα των ατόμων με αναπηρίες σε όλη τη Βόρεια Αγγλία και με τις ε, αντίστοιχες οργανώσεις που υπάρχουν. Στόχος της γνωμοδότησης είναι να ε, περιγράψει μια τολμηρή ευρωπαϊκή στρατηγική από την σκοπιά των αρμοδιοτήτων της, δικές, της δικής μας Επιτροπής. Όπως γνωρίζετε είναι περιορισμένος ο όγκος του κειμένου, το, το, του, το, μέγεθος του κειμένου, γι' αυτό και επικεντρώθηκα σε κάποια βασικά θέματα. Να λαμβάνετε υπόψη η διάσταση των ατόμων με αναπηρίες ευρωπαϊκές πολιτικής, ε, το να δοθεί προσοχή ε, σε ανθρώπους με αναπηρίες και ειδικέ εκπαιδευτικές ανάγκες από την πρώιμη και προσχολική ε, ηλικία έως και την ενηλικίεσή τους και ε, την μετάβασή τους στην απασχόληση. Εμπόδια για την κινητικότητα που παραμένουν σοβαρό εμπόδιο, ψηφιοποίηση. Το σχέδιο της γνωμοδότησης είναι αποτέλεσμα μιας πολύ καλής συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών και με εκπροσώπους των ατόμων με αναπαραγωγές απειρίες. Ε, έχουμε μιλήσει και συνεργαστεί με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την χωρίς διακρίσεις εκπαίδευση ε, και τα άτομα με αναπηρίες. Όσον αφορά την ε, ψηφιοποίηση, εγώ εκπροσώπησα την Επιτροπή Κούλτ στην IGF, όπου και μίλησα με πολλούς ανθρώπους που εργάζονται στον τομέα αυτών και έχουν αναπηρίες θέλω να συμπληρώσουμε και να βελτιώσουμε την ε, έκθεση μέσω της ε, γνωμοδότησης. Επίσης θα ασχοληθώ με ζητήματα κινητικότητας, απασχόλησης, εκπαίδευσης, ε, πρόσβαση στον αθλητισμό, ψηφιακή εποχή, συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και κοινωνική ζωή. Αυτό που μου έδωσε κίνητρο να ασχοληθώ είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι με από τον τόπο μου ε, ε, πολλές φορές εμποδίζονται ή δεν μπορούν να συμμετέχουν στην δημοκρατική διαδικασία. Γιατί πολλές φορές δεν υπάρχουν τα χρήματα. Άρα πολλές φορές είναι πολύ σημαντική και αυτή η διάσταση της ε, δημοκρατικής συμμετοχής. Όπως ε, και άλλα μέλη της Επιτροπής μας και εγώ ε, έχουμε ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα. Είμαστε υπεύθυνοι, πολλοί από εμάς, για την υλοποίηση της CRPD και κάνουμε προσπάθειες ε, προκειμένου να εξασφαλίζονται τα δικαιώματα των ατόμων με που προβλέπονται στη συνθήκη αυτή. Γι' αυτό και με μεγάλη χαρά ανέλαβα αυτή τη γνωμοδότηση, γνωμοδότηση και προσβλέπω στο να μου υποβληθούν και προτάσεις, ιδέες και από τους συναδέλφους. Ευχαριστώ πολύ Τζούλη. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους Σκιώδης. Ο κύριος Μαλτέζη είναι ο μόνος που είναι αυτή τη στιγμή εδώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την Τζούλη για την ε, δουλειά της, την οποία συμμερίζομαι απολύτως ε, και για τη θέση που πήρε. Θα ήθελα να υπενθυμίσω κάτι το οποίο αναφέρθηκε χθε και από τη Σίλβια Κώστα, γιατί εμείς ε, θα δουλέψουμε πάρα πολύ πάνω στον εξυγχρονισμό και μας απασχολεί άλλωστε ο εξυγχρονισμός της εκπαίδευσης, των συστημάτων επικοινωνίας, για την προσβασιμότητα κτλ. Έχουμε την τύχη να ζούμε σε μια εποχή που η τεχνολογία επιτέλους μας παρέχει τα εργαλεία και τον τρόπο έτσι ώστε να συμπεριλάβουμε ε, στην ζωή, ε, στην κοινωνία ανθρώπους που μέχρι τώρα ήταν αποκλεισμένοι, περιθωριοποιημένοι. Και πιστεύω ότι μια και όπως είπε και η Τζούλη ε, προηγουμένως είναι και θέμα πολιτικής, πιστεύω και μια και η αγορά, η αγορά συγγνώμη, δεν πρόκειται να το κάνει, ε, πιστεύω λέω ότι είναι ε, μια μεγάλη ευκαιρία που πρέπει να εκμεταλλευτούμε. όλοι γνωρίζουν βεβαίως ότι υπάρχουν περικοπές ε, στις, ε, στη σχολική εκπαίδευση. Ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι ε, δεν θέλουν να εγκρίνουν την προσβασιμότητα γιατί αποτελεί ένα κόστος, αν και συγκρινόμενοι με το κοινωνικό κέρδος Προφανώς δεν είναι κόστος, αλλά ε, νομίζω ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία μας δίνουν την δυνατότητα πλέον να εξυγχρονίσουμε ε, τον, ε, την εκπαίδευση στην Ευρώπη. Θα πρέπει να ξεμπλοκαριστεί η οδηγία για την προσβασιμότητα. Το κείμενο αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας το βρίσκω τέλειο. Παρά το μικρό του περιορισμένο εύρος το μόνο που έχω να πω στην Τζούλι Ward είναι ότι ίσως καλό θα ήταν ε, να γίνει μία ε, αναφορά στους ε, ανθρώπους με αναπηρία που είναι ταυτόχρονα και μετανάστες πρόσφυγες και που χρήζουν ειδική βοήθειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Σίλβια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την ε, Τζουλή για την επιμονή, την υπομονή και το πάθος ε, με το οποίο αντιμετώπισε τα θέματα τα οποία ανέφερε στην έκθεσή της. Συμφωνώ απολύτως με όλα αυτά που είπε. Τα σημαντικά θέματα τα οποία πρέπει να θυγούν στην έκθεση αυτή είναι ακριβώς αυτά τα οποία ανεφέρθησαν. Εγώ θα ήθελα όμως να υπογραμμιστεί κάτι ακόμα περισσότερο το δικαίωμα, όχι ευκαιρία, το δικαίωμα ε, των ε, ανθρώπων με αναπηρία να έχουν πρόσβαση στα σχολεία. Μετά βεβαίως μπορεί κανείς να αναφέρει όλα τα <clears throat> εργαλεία τα οποία μπορούν να υπάρξουν έτσι ώστε ε, να υποστηριχτούν και οι χώρες, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, κάποιες μορφές ειδικής παρακολούθησης ή βοήθειας αλλά νομίζω ότι είναι σαφές ότι θα πρέπει αυτός να είναι ευρωπαϊκός στόχος ε, και το ε, ζητούν ε, οι ενώσεις οι οποίες ασχολούνται με την εκπαίδευση και με τους αναπήρους. Στην Ευρώπη έχουμε αρκετή εμπειρία όσον αφορά διαφοροποιημένα σχολεία, ξεχωριστές σχολικές διαδρομές και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημείο το οποίο θα πρέπει εντόνως να υπογραμμίσουμε. Επίσης, ε, το θέμα του ε, τι γίνεται μετά την υποχρεωτική εκπαίδευση. Πολύ συχνά άτομα με αναπηρία ε, βοηθούνται μέχρι να τελειώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, αλλά τι γίνεται μετά. Και επομένως και μέσω χρήσης εργαλείων όπως είναι η blended education, όπως είναι η εξαποστάσεως ε, εκπαίδευση, θα πρέπει να ε, βοηθηθούν ε, άτομα με αναπηρία τα οποία θα συνεχίσουν και στην τετροβάθμια εκπαίδευση. Υπάρχουν και τώρα, αλλά είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι καταφέρνουν να ολοκληρώσουν και τον τριτοβάθμιο κύκλο. νομίζω λοιπόν ότι εδώ έχουμε μια καλή ευκαιρία να δούμε τον πολιτισμό όχι μονάχα σαν ε, θεατές ε, αλλά και σαν ε, πραγματικοί δρόντες εντός. Πιστεύω επίσης ότι το θέμα της ηθαγένειας είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Πριν από λίγο καιρό είχαμε την 20η επέτειο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρία. Πρέπει να σας πω με περηφάνεια ότι η Φράγκα Φαλκούτσι το 1977 άνοιξε το, το σχολείο ε, σε άτομα με αναπηρία σε ολόκληρη την Ιταλία. Μπορεί να έχουμε πολλά στραβά, αλλά γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανη. Ε, βεβαίως ε, ε, ο δρόμος δεν ήταν πάντα ανοιχτός και στρωμένος με ροδοπέταλα, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αγωνιστούμε γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σόντροβα, η οποία εκπροσωπεί και την Επιτροπή στη CRPD. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την γνωμοδότησή της. Κατανοώ ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε βεβαίως κάποια ευθύνη. Ε, ε, γίνονται προσπάθειες ένταξης των ε, των ε, ανθρώπων με αναπηρία σε εθνικό επίπεδο, αλλά νομίζω ότι όλοι περιμένουν κάποια δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, πέρσι έγινε μια δράση, ας πούμε, για τους ανθρώπους με προβλήματα ακοής σε επίπεδο ευρωπαϊκό και η Επιτροπή Πολιτισμού βεβαίως ε, ε, ασχολήθηκε ιδιαιτέρως ε, όσον αφορά το σκέλος της πρόσβασης στις οπτικοακουστικές υπηρεσίες. Οι άνθρωποι αυτοί περιμένουν η Ευρώπη να τους βοηθήσει και επομένως να δοθεί μια λύση η οποία να ξεπερνάει τα κράτη. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε με συγκεκριμένο τρόπο τους ανθρώπους ε, Ας πούμε, ε, η Julie Ward αναφέρεται στην έκθεσή της ε, στο Erasmus Plus. Ε, ενδεχομένως, ας πούμε, θα μπορούσε να υπάρξει ένα φόρουμ στο οποίο οι άνθρωποι με αναπηρία να προωθήσουν τα συμφέροντά τους μέσα στα πλαίσια του Erasmus Plus. Ευχαριστώ πολύ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλει κανείς να λάβει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Για να σας δώσω μια εισαγωγή, το Φεβρουάριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δημοσίευσε την έκθεση προόδου για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για άτομα με αναπηρία. Εκεί παρουσιάζαμε την πρόοδο που έχει επιτελεστεί από το 2016, αλλά η στρατηγική είναι μέχρι το 2020 και οι στόχοι παραμένουν ενισχύει και θα συνεχίσουμε την εφαρμογή μας. Αλλά ταυτόχρονα βρισκόμαστε το 2017 και είναι μια καλή διαδικασία. Μάλλον μια καλή ευκαιρία να αρχίσουμε τη διαδικασία προβληματισμού για το τι μέλη γενέστε μετά το 2020. Και στα πλαίσια αυτά φυσικά οι απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύτιμες. Προφανώς θα αποταθούμε και σε φορείς ετομών με αναπηρίες και θα αρχίσουμε μια διαβούλευση έτσι ώστε μέχρι το 2021 να έχουμε έτοιμη τη νέα στρατηγική. Σε ό,τι αφορά ε, την δική σας επιτροπή, την ε, εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Έχουν γίνει πολλά μέχρι τώρα, αλλά απομένουν άλλα τόσα. και θέλουμε τις απόψεις σας για το πώς θα υποστηρίξουμε καλύτερα τα κράτη-μέλη για τη συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία στην παιδεία και την αγορά εργασίας. Ε, θέλουμε να συμμετέχουν οι ευρωβουλευτές στις συνεχιζόμενες συζητήσεις για τις συνθήκη του ε, για τα υπόλοιπα κείμενα που είναι στον τριμερή διάλογο, για την προσβασιμότητα ιδιαίτερα των ηλεκτρονικών βιβλίων ε, που συμπληρώνει τη συνθήκη του Μαρακές που έχει να κάνει με τα τυπωμένα βιβλία. Καλωσορίζουμε τις προτάσεις σας και των διαφόρων εισηγητών και προσβλέπουμε σε μια συζήτηση για μια στρατηγική φιλόδοξη και χρήσιμη μετά το 2020. Ευχαριστώ πολύ. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τζούλη, θες να ξαναμιλήσεις, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση και για τις προτάσεις σας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε η Σίλβια, να τα δούμε όλα αυτά υπό το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι πολύ σημαντικό γιατί καμιά φορά τα θεωρούμε όλα αυτά δεδομένα που δεν είναι καθόλου δεδομένα και αυτονόητα. Και την ευχαριστώ για αυτό το σχόλιο. Οι αναπηρίες έχουν πολλές μορφές και πολλές αναπηρίες είναι και κρυφές και θα πρέπει μονίμως να υπενθυμίζουμε στις κυβερνήσεις και στις τοπικές κοινωνίες και στους ομολόγους μας ότι όλοι είμαστε υποψήφιοι ανάπηροι. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει σε κάποιους άλλους. Είναι μια ανθρώπινη κατάσταση ε, και αφορά ένα ποσοστό του πληθυσμού. Και καθώς μεγαλώνουμε και όλα στην ηλικία όλο και κάποιο κουσούρι λόγω θα έχουμε. Η ανάπηρη δεν είναι κάτι εκτός της ε, κοινωνίας μας. Είναι τμήμα της κοινωνίας και είναι κάτι ε, το οποίο μπορεί να μας συμβεί και εμάς μια αναπηρία. γίνεται μια πολύ ωραία καμπάνια ότι τίποτα για μας χωρίς εμάς. Είναι πολύ ωραία αυτή η εκστρατεία. Θα πρέπει όλα αυτά που λέμε και κάνουμε να είναι σε πλήρη συνεννόηση και αγαστή συνεργασία με την κοινότητα των ατόμων αναπηρία. Πολύ σωστό αυτό που είπατε για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Επισκέφτηκα το κέντρο το μεταναστών, το καταβλισμό ε, στο Καλέ και κάποιος προσπαθούσε απελπισμένα να επικοινωνήσει μαζί μου και κατάλαβα ότι ήταν κουφός. δεν ήταν απλώς στο Καλέ, στον καταβλισμό αυτό που δεν είχε τίποτα, αλλά δεν μπορούσε να επικοινωνήσει, αφγανός ήταν, ε, δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με τον κόσμο. Είχε πολλά προβλήματα. Ε, απλώς και μόνο για να κάνει μια συζήτηση, για να είναι τμήμα μια εκστρατείας που προσπαθούσαν να στήσουν εκεί. Πραγματικά με ενδιαφέρει πολύ και έχω μεγάλη ευαισθησία αυτό το θέμα των προσφύγων και των μεταναστών. Και σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σημαντικό είναι όντω να έχουμε αυτή τη ματιά με ευαισθησία ε, με κατανόηση, γιατί αναπηρία μπορεί να μας αφορά και μας. Ε, είναι το τμήμα της ζωής μας και όσο περνάει η ηλικία φυσιολογικό είναι ε, να έχουμε τέτοια φαινόμενα και εδώ βλέπουμε και στον εαυτό μας. Ευχαριστώ πολύ για την ανταλλαγή απόψεων. Θυμίζω και πάλι η προθεσμία για τις τροπολογίες 29 Ιουνίου. Έχουμε τίποτα άλλο στα διάφορα. Έχω μια ανακοίνωση να σας κάνω, γιατί σας έχω προσκαλέσει και αυτό είναι θέμα και πολιτικής ε, συμπαράστασης. Ήταν Παγκόσμια ημέρα προσφύγων και εδώ απ' έξω στην Εσπλανάτα έχουμε ένα χρυσό ε, περίπτερο. Κοντέινερ είναι βασικά. Ε, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε με πρόσφυγες. Ε, κάποιοι συνάδελφοι είπαν ότι θα πάνε. Κώστα, Βέτα, Σιλβίκη Γιόμ, Σαντιάγο φίσα και Λιάν Ροντρίγκε. Αν έχετε χρόνο, ελάτε και εσεί μαζί μα τώρα. Και είναι καλή η ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με πρόσφυγε. um, next... Επόμενη συνεδρίαση, 29 Ιουνίου, από τι 9 ω τι 12.30. Η Σίλβια Κώστα και πάλι. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Ειλικρινά για αυτή την πρωτοβουλία που με ευχαριστεί βεβαίως. Να υπενθυμίσω στους συναδέλφου, γιατί θα τους δούμε, θα βρεθούμε στις 29, ε, στις 28 όμως ε, υπάρχει μία πρωτοβουλία από πλευρά Ιταλικών Δήμων ε, για τη λεγόμενη χάρτα του Σαν που είναι ένα θαυμάσιο υπέροχο χωριό κοντά στη Σιένα. Έχει ήδη κυκλοφορήσει μεταξύ δημάρχων ε, στην Ιταλία, αλλά θέλουμε να κυκλοφορήσει και σε ολόκληρη την Ευρώπη ε, για, ε, για την υποδοχή από πλευρά των Δήμων και Κοινοτήτων της Ευρώπης, κυρίως οι ανήλικοι ασυνόδευτοι. Θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω λοιπόν αυτή την πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ. Εγώ να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς μας, ευχαριστούμε και εμείς και ολοκληρώθηκε η συνεδρία.